καλό βαθμό τις διαπραγματεύσεις σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος που στο τέλος του Δεκεμβρίου εξέφρασαν σαφέστατη υποστήριξη στα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου με 41 ψήφους υπέρ και που πιστεύω μας εμπνέουν να ψηφίσουμε και σήμερα το μεσημέρι θετικά. Έχουμε λοιπόν αναθεώρηση της οδηγίας 2001 για την, ηθελη, για την αθέλητη μάλλον διάδοση σπόρων γενετικά τροπημένων οργανισμών και αντίστοιχα τη χρήση του σε εκτρεφόμενα ζώα. Ε, το πεδίο εφαρμογής θέλω να επισημάνω ότι έχει να κάνει με την καλλιέργεια, με την ε, χρήση σε καλλιέργεια, όχι με τις εισαγωγές ούτε με τη μεταφορά. Δεν ανοίγουμε τη γενικότερη συζήτηση ως προς τη χρησιμότητα των γενετικά τροπημένων οργανισμών στη γεωργία και τη διατροφή. Και περνάω στην ουσία των συζητήσεων ε, τη ψήφου του Κοινοβουλίου και τα αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου αυτή τη τελευταία στιγμή, 3 Δεκεμβρίου, μέσα στη βαθιά νύχτα, όπου μπορέσαμε να προχωρήσουμε σημαντικά σε σχέση με τι ε, ε, αποφάσει του Συμβουλίου του Ιουλίου. Και είναι πολύ σημαντικέ οι πρόοδοι αυτοί, γιατί είχαμε μια ομόφωνη συμφωνία του Κοινοβουλίου που προωθήθηκε. Οι δύο συνομοθέτε. Ε, κατέβαλαν προσπάθειες για αμοιβές υποχωρήσεις κερδίζει πάντως το κοινοβούλιο ε, ως προς τη θέση του διότι το 2000, σε σχέση με το 2001 ένα κράτος μέλος το οποίο είναι στη μειονότητα και καλλιεργεί ε, γενετικά τροπημένους οργανισμούς πρέπει να, και υποχρεωτικά να λάβει μέτρα στην παραμεθόριο περιοχή του ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνο τη επιμέλωση. Κυρία Πρόεδρε, έχει πάρα πολύ φασαρία με στην αίθουσα. Επίση, επίσης, σε σχέση με το επίκεντρο τη οδηγία, τις περιφημε διαδικασιες διαδικασίε opt-out, αυτοεξαίρεση, με βάση τι οποίε ε, μπορεί να ε, προχωρήσει ένα κράτος μέλος που δεν θέλει να καλλιεργήσει γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Ένας νέος ρόλος αποδίδεται πλέον στην επιχείρηση που θα εφαρμόσει την νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως έχει οθετήσει το κείμενο του Συμβουλίου σε ένα βαθμό έναντι και θα σας το επιβεβαιώσουν οι σκιώδεις συγγητές. Ελείψει λοιπόν η ασδήποτε διάθεση για υποχώρηση από το Συμβούλιο. Ωστόσο έχουμε πολύ σημαντικά κέρδη εξασφαλίσει Κοινοβούλιο την ε, άρση της αιρεσιμότητας στη φάση 1 και τη φάση 2, δηλαδή υπάρχουν δύο μπαλαντέρ θα λέγαμε, δύο περιθώρια ευκαιρίας για να περιοριστεί αυτή η καλλιέργεια στην επικράτη ενός κράτους. Μπορεί να, συν, να συναδιαλλαγεί με την επιχείρηση που πολλοί τους σπόρους, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να το πράξει το κράτος αυτό και έχει, όπως όριζε το Συμβούλιο στις προτάσεις του, και επίσης έχει δέκα χρόνια στη διάθεσή του και όχι δύο μόνο, για να προχωρήσει στη δεύτερη φάση με έναν ανοιχτό κατάλογο ε, αιτιολογιών όπως προστασία της βιοποικιλότητας του περιβάλλοντος και άλλα πολλά και επίσης το Συμβούλιο υποχώρησε και δέχθηκε να επεκτείνει την προστασία στις ομάδες γενετικά τροπημένων οργανισμών. Ναι, Πρόεδρε, παίρνω από τον χρόνο που θα είχα ως δευτερολογία και συνεχίζω. Και εδώ, απευθυνόμενοι στους ε, αναποφάσεις τους, θα πω ότι δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική σε αυτή την συμφωνία. Δεν είναι δυνατό να δεχθούμε ως επιλογή ρεαλιστική το καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή το status quo εκτός και αν θέλουμε την ζούγκλα, την απόλυτη απορρίθμιση και την επικράτηση του ισχυροτέρου. Νομίζω ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή μπορούμε να πιέσουμε τον, τον πρόεδρο Γιούνκερ να προχωρήσει τη μεταρρύθμιση, να προχωρήσει τη ρύθμιση των γενετικά τροπημένων οργανισμών, να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα μέσα να κάνουν σεβαστές τις θεμητές επιλογές τους με την νομοθεσία αυτή, χάρη στην νομοθεσία αυτή προχωρούμε, εισακούμε και προωθούμε τις επιλογές των κρατών μελών. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Συγγετρία και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Αντρουκάητης, εξ ονόμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Madam President, honorable members. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σας σήμερα το πρωί Χρειάστηκε πολύ καιρό, μία πενταετία περίπου, αλλά έχουμε φτάσει στο τέλος αυτή τη διαδρομή. Τότε δεν θα σκεφτόμουν ποτέ ότι θα είχα αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ μετά από μια επιτυχημένη δεύτερη ανάγνωση θέλω να συγχαρώ την κυρία Φεντερικρή στην εισηγήτρια για την αποτελεσματική της καθοδήγηση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους κοινούς εισηγητές για την υποστήριξή τους. Αυτές οι συλλογικές λοιπόν προσπάθειες μας βοήθησαν να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτό το έργο. Επιτρέψτε μου να σας ε, θυμίσω το ιστορικό. Σήμερα ένα μόνο είδος επιτρέπεται να καλλιεργείται στα κράτη-μέλη. Πέντε κράτη-μέλη το καλλιεργούν. Εννέα κράτη έχουν ε, λάβει μέτρα για να ε, αποτρέψουν ε, την καλλιέργεια στην επικράτειά τους. Αυτά τα μέτρα όμως δεν θεωρήθηκαν αιτιολογημένα από την ΕΦΣΑ. Και τώρα είναι στα χέρια των εθνικών δικαστών που έρχονται και τα ακυρώνουν. Δηλαδή, χώρε που θέλουν να απαγορεύσουν τι καλλιέργειε μεταλλαγμένων στην επικράτειά του δεν επιτρέπεται να το κάνουν λόγω τη κείμενη νομοθεσία ε, που δεν επιτρέπει στα κράτη-μέλη να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των λαών τους και ε, την κείμενη νομοθεσία. Αυτό δημιουργεί τεράστιες εντάσεις ανάμεσα ε, στο νόμο, το κοινό και τα κράτη. Και επίση οι εταιρείε θεωρούν ότι παραμελούμε τα συμφέροντά του και μειώνεται η αξιοπιστία όλων που ενέχονται σε αυτή την προσπάθεια εκτίμηση κινδύνου για ε, τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΦΣΑ και τέτοια για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό μέχρι το 2009 13 ε, κράτη-μέλη ζήτησαν μια λύση να δοθεί. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή έκανε μια λογική πρόταση το 2010 απαντώντας αυτή την έκκληση. Είναι διπλή στόχη. Ο πρώτος, να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα έγκρισης με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και ενιαία ασφάλεια ομοιόμορφη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δεύτερος στόχος ήταν να αναγνωρίσουμε σε πλήρη σεβασμό των συνθήκων την ελευθερία κάθε κράτους μέλους να αποφασίζει ελεύθερα εάν θα επιτρέψει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή όχι. Ναι στο έδαφο του. Και χαίρομαι που το παρόν κείμενο σήμερα ε, ανταποκρίνεται πλήρω και στου δύο στόχου. Θα έχουν τον τελικό λόγο τα κράτη-μέλη ως προς την καλλιέργεια, ανάλογα με την εθνική κατάσταση του καθενό. Υπάρχουν χώρε που ήδη καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Εκείνε που θέλουν να περιορίσουν ή ακόμα και να απαγορεύσουν επίση δίνονται να το πράξουν. Η ε, ελεύθερη επιλογή είναι εξασφαλισμένη και οι χώρε που ήδη καλλιεργούν θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποτραπεί η διασυνοριακή μετάδοση επιμόλυνση σε μια γειτονική χώρα. Επίσης, ε, προσεχώς θα αναβαθμιστεί και θα επικυρωποιηθεί ε, ο τρόπος με τον οποίο εκτιμούμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα ήθελα να τονίσω ότι τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση πάντα και ακόμα να ε, λαμβάνουν τα μέτρα που εκείνα θεωρούν σωστά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Αν υπερψηφίσετε αυτή την νομοθετική πρόταση για την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών, θα δώσετε στα κράτη-μέλη νομική ασφάλεια με ε, στιβαρά εργαλεία για να μπορούν να αποφασίζουν ε, ήδη από φέτος, από την άνοιξη του 2015. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανειλημμένα εκλήθη να κάνει περισσότερα για να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών και σας εγγυώμαι ότι αυτή η νομοθεσία απαντά σε αυτή την έκκληση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα ήθελα να κάνω την εξή δήλωση. Όταν ακολουθεί τη διαδικασία ε, αδειοδότησης, η Άγκριση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σεβαστεί πλήρως και θα σέβεται πάντα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Μεταξύ αυτών είναι και η δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν πλήρω την καλλιέργεια ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφος. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you. Now we move to... Και εμεί ευχαριστούμε. Και τώρα οι ομιλητέ εξ των πολιτικών ομάδων. κυρία Κώστιγκερ πρώτα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Μετά από τέσσερις μήνες σκληρής δουλειάς επιτέλους καταφέραμε να φέρουμε στην Ολομέλεια μία πρόταση για την οποία έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά την αυτοδιάθεση και την ε, ε, αυτόνομη απόφαση των κρατών μελών. Μετά από πολλά χρόνια το καταφέραμε και πραγματικά θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Ρίζ, μεταξύ όλων και για την επικοδομητική συνεργασία. Το νομικό κείμενο είναι μεγάλη πρόοδο προ μεγαλύτερη αυτοδιάθεση και μεγαλύτερη επικουρικότητα. Και στο εσωτερικό των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντίσταση κατά τη γενετική τεχνολογία το Pioneer 1507. Θυμάστε τι έγινε. 19 κράτη-μέλη ήταν αντίθετα με την έγκρισή του. Αυτό είναι γεγονός το οποίο δεν ε, μπορούμε να παραβλεψουμε 8 Οχτώ κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν αρχίσει και καλλιεργούν τον το μόν 810 ε, μάλλον ε, τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη έχουν απαγορεύσει την καλλιέργεια του μόνο 810 βάσει τη ρήτρα προστασία, όπω ονομάζεται. Ε, ενώ κάποιε άλλε καλλιεργούν. Είναι μια κατάσταση λοιπόν αυτή αβίωτη, αφόρητη και θα πρέπει να δοθεί ένα τέρμα. Ε, προβλέπεται τώρα μια διαδικασία δύο φάσεων και έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή νομική ασφάλεια σεβόμενη πάντα και ενισχύοντας την τα Ξέρω ότι δεν είναι το απάβγασμα της σοφίας, αλλά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η πρόταση και παρακαλώ τους συναδέλφους να την υπερψηφίσουν. Speaker is, uh... Τώρα, κύριος Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα αν απαγορέψει ένα κράτος μέλος την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ε, σέρνεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατόπιν ε, μήνυσης της Μονσάντο. Η τελευταία συμφωνία όμως του Μερή Διάλογου αλλάζει τα πράγματα. Είναι σημαντικό να το πούμε. Χωρίς τη συμφωνία αυτή θα, θα παρέμεναν τα πράγματα όσοι είχαν, δηλαδή θα μπορούσε ένα κράτος μέλος να δεχτεί την καλλιέργεια τροποποιημένων οργανισμών λόγω έλλειψης θέσης του Συμβουλίου. Η Γαλλία θέλει να απαγορεύσει τα τροποποιημένα και σε αυτήν την μακρά συζήτηση και διαπραγμάτευση με ένα Συμβούλιο που καθυστερεί συνεχώς μπορέσαμε με τον κύριο Ρίζ να ενισχύσουμε την, την να ενισχύσουμε την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία αυτή όντως δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στα κράτη-μέλη που αντιτίθενται στην καλλιέργεια τροποποιημένων οργανισμών. Η απαγόρευση θα επιτρέπεται για λόγους αγροτικούς, περιβαλλοντολογικούς και οικονομικούς είναι περισσότερη ασφάλεια για τους γεωργούς παραδοσιακών καλλιεργειών. Σε δύο χρόνια τα κράτη-μέλη μπορούν να πάρουν μέτρα για να εμποδίσουν για να απαγορεύσουν την παρεμπόδιση των παραδοσιακών καλλιεργειών υπέρ των τροποποιημένων. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και για τους καταναλωτές. Η Κομισιόν ανέλαβε τη δέσμευση να κάνει την αποτίμηση του κινδύνου, την αξιολόγηση μέσα σε δύο χρόνια από τώρα. Άλλη νίκη για τους καταναλωτές. Πείσαμε την Κομισιόν να μην δώσει καμία νέα άδεια για καλλιέργεια τροποποιημένων πριν αρχίσει να ισχύει αυτή η οδηγία. Επρόκειτο για αγώνα δύσκολο, αλλά νομίζω ότι τον κερδίσαμε. φεύγει η αυτή δεν είναι παρά μια αρχή πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας κατά των τροποποιημένων. Thank you, uh, Mrs. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέρλινγκ δύο λεπτά. Νομίζω ότι η προτινόμενη συμφωνία αντικατοπτρίζει τις επιλογές των κρατών μελών για το αν θα καλλιεργήσουν ή όχι γενετικά τροποποιημένα ε, η διαδικασία αυτή στην ουσία τεκμηριώνει την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αδειοδοτεί ε, στη συνέχεια των αιτήσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί γιατί της λείπει το πολιτικό θάρρος. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καθορίζονται από τη συνθήκη στον συγκεκριμένο τομέα δεν είναι απόλυτες και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και στους επόμενους τομείς. Ε, βέβαια ο διάβολος βρίσκεται ή κρύβεται στις λεπτομέρειες. Η συμφωνία θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν άμεσα και σε εθνικό επίπεδο στην αδειοδότηση. Θα επιτρέψει, θα έλεγα, στις εθνικές υπηρεσίες να αδειοδοτούν ομάδες γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών και όχι με μονομένα φυτά όπως μέχρι τώρα. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τις διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν δοθεί η τελική άδεια κυκλοφορίας. Συνεπώς θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε οι προτινόμενες λύσεις να μην υπονομευθούν από την ισχύουσα ήδη κοινοτική νομοθεσία υπάρχει μια δυσανάλογη δαιμονοποίηση των γενετικά τροποποιημένων. Τα κράτη-μέλη στην ουσία κλείνουν την πόρτα στην μικρότερη χρήση υδάτινων πόρων, στη μεγαλύτερη παραγωγικότητα και στα υγιέστερα προϊόντα, κάτι το οποίο θα έχει συνολικότερα ευεργετικές συνέπειες στον τομέα της υγείας. Οι αδειοδοτήσεις λοιπόν ελπίζω να δοθούν τα κράτη-μέλη που θέλουν να αναπτυχθεί η Ευρωπαϊκή Γεωργία σαν οι καλύτεροι στον κόσμο ε, περιμένουν να μπορέσουν να στραφούν ξανά στο δρόμο της πρόοδου.